με βάση το άρθρο 69C παράγραφος 1 του εσωτερικού κανονισμού. Οι εκθέσεις οι οποίες αποτελούν εντολή για αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και οι τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της Ολομέλειας. Με βάση το άρθρο 69C παράγραφος 2 ένα αριθμός ε, πολιτικών, ε, συγκεκριμένων πολιτικών ομάδων μπορούν να ζητήσουν γραπτός μέχρι ε, αύριο, 3η, 24 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Εάν δεν υπάρξει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για την απόφαση να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι, οι επιτροπές αυτές μπορούν να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις. Με βάση το 6 του κανονισμού, ο πρόεδρος τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με ενημέρωσε